μπορέσουμε όλοι να πούμε ότι ήταν αντικειμενική αυτή η έκθεση, ότι ήταν αντικειμενικές αυτές οι εκθέσεις και ότι αντανακλούσαν, αντικατόπτυσαν την κατάσταση στην περιοχή αυτή του κόσμου αντικειμενικά. Πρόεδρο, ευχαριστούμε συνάδελφε Φορέμπα. Η κοινή συζήτηση εδώ ολοκληρώθηκε. Η ψήφιση των δύο εκθέσεων θα διεξαχθεί αύριο στις 11 και 30. Επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού, σύμφωνα με το άρθρο 150 του κανονισμού. Και πρώτα απ' όλα η κυρία Ζαμπόσκα θα παρέμβει. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το μεσημέρι έγινε ευρύτερα λόγο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και υπό αυτό το πρίσμα δύο στοιχεία. Τον Απρίλιο 2012 κάνουμε λόγο για τα δικαιώματα του ανθρώπου παγκόσμια και για τα δικαιώματα του ανθρώπου ε, για, το έτος 2010 και κάποια πράγματα τα οποία όταν ε, έχουμε τέτοια θέματα ε, πολλές φορές ε, αντανακλούν μια τοποθέτηση κάποιου φοιτητή που ενασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτή η έκθεση το 2011 δημοσιεύτηκε και ασχολούμεθα με αυτή σήμερα. Για τη Λευκορωσία, το καθεστώς Λουκασένκα το 2010 μετεξελίχθηκε προς το χειρότερο, με, την χειρότερο, με το χειρότερο πρόσωπό του. Και γι' αυτό η το παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκεϊ δεν θα θέλαμε να διεξαχθεί στην ε, Λευκορωσία. Η ομάδα της Λευκορωσίας αξίζει μια τέτοια εκδήλωση. Όμως το καθεστώς Λουκασέρκα δεν πρέπει να καταχραστεί μια τέτοια ευκαιρία, μια τέτοια εκδήλωση, αν εμείς αποδεχθούμε να διεξαχθεί εκεί αυτό το πρωτάθλημα. Ο συνάδελφος Μίσκι δεν είναι παρόν και γι' αυτό θα λάβει τον λόγο η συνάδελφο ε, Μπιλμπάου Μπαράντικα τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Στις 26 Αυριλίου θα έχουμε την 25η ε, επέτειο του βομβαρδισμού της Γκουέρνικα. Μαζική επιθετικότητα κατά αμάχων. Κάτι το οποίο συνεχίστηκε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Φράγκο έκανε το ίδιο κατά της βασικής ε, ταυτότητας. Ήταν βασικός στόχος της δικτατορίας. Και όμως έτσι χτυπήθηκε αυτό το σύμβολο της ε, της ειρήνης με αυτόν τον πίνακα του Πικάζου. Και ε, σήμερα έχουμε κάποιους αναθεωρητές της ακροδεξιάς που θεωρούν ότι ε, με τα, με το μετασυμβολικό ισπανικό στηρίχθηκε πάνω σε αυτήν την ατιμορρησία του φραγκισμού. Οπότε με αυτήν την επέτειο της, του βομβαρδισμού της Γκουέρνικα θα πρέπει να ζητήσουμε που των θυμάτων γιατί περάσανε τόσα χρόνια και θα πρέπει ομένω να κάνουμε αυτό το οποίο δεν έκανε ο φραγκισμός ε, που έπληξε και ζημίωσε τόσα εκατομμύρια προσώπων. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Μπιμπάου Μπαράντικα. Αφόνση δεν παρίσταται δυστυχώς. Ο κύριος Μιγκάσκι λοιπόν έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αναφερθώ στα όσα είπε η κυρία Ζαμπόρσκα και να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου. Το δικτατορικό καθεστώς Λουκασένκα στην Λευκορωσία, στην Πελαρούς. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε και δύο κρατούμενους που απελευθερώθηκαν. Είναι ένα θετικό στοιχείο αυτή η απελευθέρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι αναμφίσιμα τοποθετείται και το καθεστώς της ε, Λευκορωσίας ε, το αξιολογεί χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Είναι θετικά αυτά τα βήματα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν περαιτέρω κρατούμενοι στις φυλακές ε, και αυτοί πρέπει να απελευθερωθούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάποιες φορές αδυναμίες. Γίνονται κάποια βήματα προς τα εμπρός και μετά βήματα προς τα πίσω, οπισθοχωρούμε. Δύο βήματα εμπρός, δύο, τρία βήματα πίσω. Γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε την υποστήριξή μας υπέρ των Λευκορώσων. Ευχαριστώ. Μουγκάνσκι τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τις τελευταίες εβδομάδες συνέβησαν κάποια επεισόδια που θα περιοριστώ ότι θα τα πω παράξενα όμως αντιπροσωπεύουν μια ιδέα πάρα πολύ σοβαρή και επικίνδυνη. Στην Ιταλία μια ομάδα ψευδοερευνητών που είναι αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο έρεσαν την πρόθεση να θέλουν να επανεξετάσουν ή να εγκαταλείψουν την ανάγνωση της θεία Κομμωδίας. Το έργο του, του Ντάντε που εξήμισαν επί αιώνες εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Το αριστούργημά του. Το πόημα παρουσιάζει, είπαν, πολλές ρατσιστικές αναφορές, αντισημητικέ και ισλαμοφοβικέ. και θα πρέπει να αναθεωρηθεί από ένα πολιτικό μάτι σωστό και μοντέρνο. Η Ένωση Αποκατάσταση των Πολιτών ζήτησε να απαγορευτούν κάποια, κάποια πιάτα να αλλάξουν ονόματα, όπως είναι το μαύρο ψωμί, παραδείγματο χάρη το το ψωμί του νέγρου γιατί είναι ρατσιστικά. Όμω αυτό είναι ένα διάχυτο συνέστημα που κρατεί στην Ευρώπη. Είναι σαν να θέλουμε να αρνηθούμε τι ρίζε μα για να ευχαριστήσουμε διάφορε ε, πολι... ε, πολιτισμού. Αλλά ένα δέντρο χωρί ρίζε πεθαίνει. Θα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση η Ευρώπη, θα πρέπει να προστατεύσει τι ρίζε τη και το παρελθόν τη. Σα ευχαριστούμε, συνάδελφε Μοργκάντη. ο συνάδελφος Μάτια, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Πορτογαλία την προηγούμενη εβδομάδα είχε ένα τελεσίγραφο το οποίο επευλήθη δημοσιονομικά που δεν ε, έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η θετική ψήφος ε, των κυβερνητικών κομμάτων δείχνει, αντανακλά την πολιτική δεκαετιών ε, ηλικιότητας και ανθρώπων που δεν σκέφτονται καν το τι πρέπει να γίνει. Η θέση των σοσιαλιστών και σε σχέση του ΠΕΔΕΣ δείχνουν, δείχνει την ανεύθυνη στάση. Αυτό καθιστά την Βουλή Βουλή στην Πορτογαλία την πρώτη βουλή που δέχεται την ταπείνωση, αποδέχεται την ταπείνωση και απεμπολεί τις ε, αρμοδιότητες της ε, η Βουλή για το αξίωμα στο οποίο εξελέγει. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήγμα αυτό. Βλέπουμε ότι η εξουσία του χρήματος ε, ξεπερνά την έκφραση της ψήφου των πολιτών. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την πολιτική αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μάτια. Ο συνάδελφος Όμπερ Μάιερ ε, είναι εδώ. Γι' αυτό ο συνάδελφο Ριβελίνη θα λάβει το. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ιταλία είναι δραματική. Η δική μα συμμετοχή στην Ευρώπη περνάει κρίση. Αυτό διότι οι Ιταλοί οι εργαζόμενοι δεν κατανοούν την Ευρώπη όταν χάνουν τη δουλειά του, διότι μεγάλε επιχειρήσει κλείνουν σε εμά και πηγαίνουν σε ευρωπαϊκέ χώρε που έχουν κόστος εργατικό χαμηλότερο. Δεν καταλαβαίνουν την Ευρώπη αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί τι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσει, αλλά αντί να το κάνει αυτό μόνο τα μεγάλε τράπεζε δεν καταλαβαίνουν την Ευρώπη όταν διώχνεται δημοκρατικά εκλεγμένη από του Ιταλού κυβέρνηση για να αντικατασταθεί από τεχνοκράτε, που μόνο λύσει στην κρίση προτείνουν την αύξηση των φόρων του καυσίμων, τη βενζίνη. Δεν καταλαβαίνουν την Ευρώπη Ευρώπη. Αν η Ιταλία αλληλεί στα σύνορα με την Κροατία, ε, πρέπει να υποστούν κανόνες που οι Κροάτες δεν σέβονται που θα μπουν σε λίγο στην κοινή αγορά. Δεν καταλαβαίνουν την Ευρώπη αν εκμεταλλεύονται τους πόρους μας χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την παλιά Ήπειρο. Όπου ε, δεν σέβονται λοιπόν την ιστορία Λοιπόν, η Ευρώπη πρέπει να σεβαστούν τα όρια της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Ριβελίνη. Ο συνάδελφος εντιού παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα της, των κέντρων κράτησης στην Ευρώπη είναι σημαντικό ζήτημα για την Ευρωβουλή ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το ενδιαφέρον ε, για αυτή την πτυχή και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας όμως δεν μπορεί να, είναι, να έχει ανώτερη προτεραιότητα από την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε ότι επανειλημμένα κατηγορούνται κάποιες χώρες ε, χωρίς κάποια τεκμήρια. Η Ρουμανία κατηγορείται επανειλημμένα για το ότι είχε τέτοια κέντρα κράτησης στη CIA και η μόνη απόδειξη εντός εισαγωγικών ή το μόνο τεκμήριο ήταν κάποια δημοσιεύματα εφημερίδων. Οι διακριβώσεις και οι ανακρίσεις ε, δεν κατέδειξαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την πτυχή των κέντρων κράτησης. Για τα, ε, τις φυλακές της CIA δεν είναι όλες οι κατηγορίες σωστές ε, και αντικειμενικές. Πρέπει να βασίζονται σε τεκμήρια και αποδείξεις Στη, Ρουμανία δεν υπήρξαν τέτοια κέντρα, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφε Έντσιο. Ο κύριος Γκάλαγκερ ακολουθεί παρακαλώ. Εγώ, Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα πρέπει με αυτά τα μέτρα της φορολογικής πολιτικής να βοηθήσουμε την Ιρλανδική οικονομία. Και έτσι θα πρέπει να έχουμε νέους νόμους για να ρυθμίσουμε τη χρηματοπιστωτική αγορά. Με τη νέα συμφωνία θα έχουμε περισσότερη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Και έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην οικονομική ανάκαμψη. με την οικονομική σταθερότητα. Επίση, θα έχουμε τι προποθέσει για δημιουργία θέσεων εργασία. Οι χώρε οι οποίε θα ακυρώσουν την συνθήκη θα μπορέσουν να καλυφθούν από τον ε, μηχανισμό σταθερότητα. Γιατί δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στι αγορέ. Όσοι είναι καλέ καινούριε συνθήκε, θα πρέπει να μα αποδείξουν το πώ σε αντίθεση περίπτωση θα μπορούν να αγορέ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Γκάλαγκερ. Ακολουθεί ο συνάδελφος Ταβάρες παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μια θλιβερή πραγματικότητα στη Γινέα Μπισάου. Για άλλη μια φορά οι στρατιωτικοί που υποτίθεται ότι θα υπεράσπιζαν την πατρίδα, το καθεστώς και το σύνταγμα επιτίθενται εναντίον όλων. Ε, σε σχέση με την έκθεση του 2008 όταν είχαμε το θέμα των ε, ε νήσων στη Γινέα Μπισάου, ακατοίκητων νήσων που θα, τις χρησιμοποιούσαν συμμορίες για το ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αυτό το οποίο συνέβη από το 2008 τι ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση απέσυρε την αποστολή στη Γινέα Μπισάου για την συνεργασία με το ίδιο το καθεστώς και τους στρατιωτικούς. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σφάλμα. Ε, είχαμε μέσα σε πολύ μικρό ε, διάστημα σημαντικότατο πρόβλημα. Κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί με επιπτώσεις σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων ε, που αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ελπίδα που θα ανοίξει για τον λαό της Γινέα Μπισάου. Θέλει να αποκαταστήσει τη ζωή του ο λαός αυτός και πρέπει να υπάρξει ελπίδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Ταβάρες. Ο συνάδελφος Σαρνέτσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πριν από δύο χρόνια ένα πολωνικό αεροπλάνο συνετρίβει και υπήρξαν πάμπολα θύματα αυτό το αεροπλάνο μετέφερε όχι μόνο τον ίδιο τον πρόεδρο της ε, Πολωνίας αλλά και τους ανώτατους αξιωματούχους, ε, τους ανώτατους ε, ηγέτες. Εδώ και αυτά τα ε, δύο χρόνια βρίσκεται, βρίσκονται τα συντρίμια αυτά, ε, αυτού του αεροπλάνου στη Ρωσία. Δεν έχουν επιστραφεί στην Πολωνία και το, το μαύρο κουτί black box δεν έχει παραδοθεί στους Πολωνίους, στις πολωνικές αρχές. Είναι ασύλληπτο, είναι αδιανόητο ότι τον 21ο αιώνα ε, δεν, ο λόγος για αυτή την τραγική, την, την καταστροφή, αυτή, αυτό το τραγικό συμβάν δεν μπορεί να διαφωτιστεί και να δούμε το τι συνέβη. Ελπίζουμε ότι θα υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Πάτων παρακαλώ. Uh, Κάποιες θέσεις εργασίας μπορούσαν να έχουν διασωθεί στο Λονδίνο. Όμω λόγω τη κοινωνική Νομοθεσία χάθηκαν και έχουμε το εργοστάσιο τη Ζάχαρη το οποίο απέλησε 30 πρόσωπα. Και αυτό διότι σήμερα με τι ποσοστώσει της δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί η ακατρέφτη ζάχαρη. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η νομοθεσία και να μπορούμε να αποθεθούμε στην στις 14 Μαρτίου μίλησα με τον Επίτροπο και του είπα ότι θα πρέπει να βοηθήσει αυτή την επιχείρηση ώστε να επιλύσει το πρόβλημά της. Μέχρι σήμερα όμως δεν μου έχει απαντήσει ο Επίτροπος και δεν είναι δυνατόν ε, σε ένα τόσο φτωχό κομμάτι του Λονδίνου να μην κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να βοηθήσει η Επιτροπή και να καταλήξουμε σε κάποια λύση σύντομα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Μπάτεν, Σέντεγκάρτ παρακαλώ. Τάκ. Ε, øh, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς τον Πρόεδρο. Εδώ και 39-40 ε, μέρες ξεκίνησε απεργία πείνας στο Μπαχρέιν ε, διαμαρτυρώμενος κατά της δικτατορίας του βασιλικού καθεστώτος και της ε, σύλληψής του. Τι έκανε αυτός ο αντιφρονών ποιο έγκλημα είναι εκείνο το οποίο τον οδήγησε στη φυλακή. Όχι βέβαια με βία, αλλά με τις δηλώσεις του και με την ειρηνική του δράση και διαδηλώσει και, και ε, διαμαρτυρία. Μετά από τόσες μέρες απεργίας πείνας ε, βρίσκεται ε, πολύ κοντά στο θάνατο. Δεν πρέπει να αφήσουμε να πεθάνει. Γι' αυτό ζητώ από τον Πρόεδρο να διασφαλίσει ότι από την ίδια την Ευρώπη θα απευθυνθεί έτοιμα αίτημα κατεπηγόντως προς τον ε, βασιλέα του ε, Μπαχρέιν ώστε να απελευθερωθεί ο κρατούμενος αυτός διότι αύριο θα είναι ήδη πολύ αργά και θα έχει πεθάνει. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Σέντεργαρντ. Ο συνάδελφος Κέλλη παρακαλώ έχει τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει και πολλού εκπροσώπους της και πολλού συναδέλφου των Φιλ Πέντεργκραπ του Σοσιαλιστικού κόμματο. Ένα Ιρλανδό πολίτη δολοφονήθηκε από τι Βολιβιανέ αρχέ εδώ και τρία χρόνια. Και φαίνεται ότι ο Μάικλ Ντουάιρ ήταν άοπλος και όμω πυροβολήθηκε στην καρδιά και τρει φορέ στην πλάτη από τι Βολιβιανέ αρχέ. Η οικογένεια φυσικά θέλει απαντήσει σε διάφορε ερωτήσει, αλλά παρά τρία χρόνια που πέρασαν, οι βολβιανέ αρχέ δεν είναι πρόθυμε να διεξαγάγουν ανοιχτή διεθνή έρευνα για το συμβάν. Ήταν εδώ ο Μάρτιν και η Κάρολαν και αδελφή η Άσλιν, και του άκουσε η Λέδη Άστον που υποστηρίζει το διάβημα αυτό. Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη ανοιχτή έρευνα 204 εκατομμύρια βοήθεια δίνουμε στη Βολιβία. Και αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να του υποχρεώσει να διερευνήσουν αυτή την, ε, να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, να επιτρέψουν την έρευνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Κέλλη. Η κυρία Κοστέλο, η συνάδελφος κυρία Κοστέλο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σαν μέλος της Task Force του Βορειού Δουβλίνου έλαβα πολλές αναφορές για βία, παρενόχληση, πιέσεις κατά οικογενειών και ηλικιωμένων γονέων χρηστών ναρκωτικών για χρέη για ναρκωτικά πολύ συχνά που συνεπάγονται πάρα πολύ μικρά ποσά. Το 2008 ε, ε ξεκίνησε μια προσπάθεια στην Ιρλανδία για να δώσει εμπιστευτικέ ε, πληροφορίε όσον αφορά το εμπόριο ναρκωτικών. Πάνω από 9.000 κλήσει δέχτηκε το κέρδο. 2.500 αναφορέ στέθηκαν στην ε, μονάδα ναρκωτικών τη Ιρλανδική αστυνομία. Θα ήθελα να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει μια κοινή προσπάθεια ευρωπαϊκή για να σταματήσουν οι απειλέ σχετικέ με τα ναρκωτικά και να είναι αριθμοί αντίστοιχοι με την απώλεια παιδιών, θύματα ατυχημάτων ε, και ιατρικά κατεπήγοντα περιστατικά. Και παρ' την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει να χρηματοδοτήσει αυτή την πολύ καλή δημόσια υπηρεσία όσον αφορά το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Ενώσεω, το πρόγραμμα Δάφνη και παρόμοιε πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα σε διεθνέ ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Κοστέλο. Ο συνάδελφος Τερμόσα Ιμπάσε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χτες γράφτηκε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των εθνικοποίησεων. Η Αργεντινή εθνικοποίησε την EPF η εταιρεία που ερχόταν από την Ερεψόλη, ήταν μονομένη σε αυτή την κίνηση και έτσι η κυβέρνηση τη Αργεντινή έγινε ο βασικότερο μέτοχο σε αυτή την εταιρεία και απέκτησε το 51% των μετοχών. Και η ρεψόλ τώρα έχει το 57% το οποίο είχε. Επρόκειτο για κάποια επίθεση στο κράτος δικαίου, έτσι δημιούργησε ανασφάλεια, έτσι υπενόμευσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Πρόκειται για μια πράξη που ήρθε πιο κοντά η χώρα στη Βενεζουέλα ή στην Κούβα. Απομακρύνθηκε από, την, από το πρότυπο της ε, πετυχημένης Βραζιλίας. Οπότε εμείς έχουμε ζητήσει από το Συμβούλιο να στηρίξει την Ρεψόλ και τους άλλους ε, επενδυτές ε, της Ευρώπης. Και έτσι θα πρέπει οι εμπορικές συμφωνίες να παγώσουν και με κάποιους μηχανισμούς να εξασφαλίσουμε ότι τέτοια πράγματα δεν θα ξαναγίνουν. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Τρεμόζα η Ο κύριος Χρυσόγελος έχει τον λόγο παρακαλώ. με αφορμή την ε, σημερινή παγκόσμια μέρα μία των εξοπλισμών ε, θα πρέπει να διδαχτούμε από τα λάθη τα οποία έκανε η ελλάδα στα θέματα αυτά από το 1974 στο 2011 η Ελλάδα δαπάνησε γύρω στα 218 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμυντικά και εξοπλιστικά προγράμματα. Μάλιστα την περίοδο 2001-2011 και παρά τη μείωση των αμυντικών εξοπλιστικών δαπανών το 2011 λόγω της μεσονομικής προσαρμογής η Ελλάδα υπήρξε ο πέμπτος μεγαλύτερο εισαγωγέας όπλων στρατιωτικού εξοπλισμού με 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια στον κόσμο μετά την Κίνα, την Ινδία, την Νότια Κορέα και τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα. Ε, Όμω και την πενταετία 2007-2011 η Ελλάδα ήταν ο μεγαλύτερο παραλήπτη γερμανικών και ο δεύτερο μεγαλύτερο παραλήπτη γαλλικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Πρέπει σίγουρα να διδαχτούμε από τα λάθη γιατί κυρίω οι μεγάλε βιομηχα... πολεμικέ βιομηχανίε υποφελήθηκαν από τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και στελέχη τη ελληνική δίκη και έλληνε πολιτικοί που είχαν την ευθύνη για την επιλογή διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αποκορύφημα είναι βέβαια η σύλληψη του πρώην Υπουργού Ελλάδα, του κ. Τσοχατζόπουλου. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Χρυσόγελε. Ακολουθεί ο συνάδελφος Βοζόβιτ. Παρακαλώ. Μικρό. Μικρόφωνο παρακαλώ. Με μικρόφωνο συνάδελφε. E, Ευχαριστώ πολύ. Ε, τελειώνει, έγινε συζήτηση για τι συμφωνίε με την Αρμενία, το Τζερμπαϊτζάν κλπ. Συζητήσαμε αυτό το θέμα. Όμως όλες οι ευρωβουλευτέ ανησυχούν και για το Ιράν, ε, που είναι κοντινό στην περιοχή. Ε, σε μέση βάση, στη Σύνοδο Κορυφής της Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να συζητηθεί το πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν Ανησυχώ ότι υπήρξε μεγάλη συγκέντρωση, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στα σύνορα με του Καυκάσου ρωσικών δυνάμεων. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να μην εμπλουτίσει άλλο ουράνιο το Ιράν, για λόγους μη ε, πολιτικούς ή ιατρικούς. Δεν θα πληροφορούμε τη Ρωσία, που συγκεντρώνε, ενώ συγκεντρωνόμαστε μόνο στο Ιράν και θέλει η Ρωσία να επανακτήσει τον έλεγχο στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστούμε συνάδελφε Βλόσοβιτς. Ο συνάδελφος Βαρκόφσκι δεν παρίσταται. Ο συνάδελφος Βάτιμο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι αυτή την εβδομάδα εις Ουάσιγκτον πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και διαφόρων πολιτικών κομμάτων του κόσμου συναντούν για να ζητήσουν τον πρόεδρο Ομπάμα μια πράξη δικαιοσύνη να ξαναδώσει την ελευθερία σε πέντε κουβανού που συνελήφθησαν το 1998 στη Φλόριδα και κατηγορούνται από την Αμερικανική κυβέρνηση για κατασκοπία και δίσδυση στη ΣΥΠΑ ω μυστικοί πράκτορε ενό ξένου κράτου, χωρί τίποτα από όλα αυτά να έχει αποδειχθεί ποτέ. Ε, υπήρξε μεγάλο κρίμα εχθρότητα στο Μαϊάμι και καταδικάστηκαν σε υπερβολικές ποινέ. παραδιάστηκαν οι διεθνεί συνθήκε όσον αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Ο ΙΕ δήλωσε ότι ήταν άκυρη αυτή η διαδικασία, αυτή η δίκη, διότι δεν υπήρχαν τα ελάχιστα χέρια για την υπεράσπιση και θα έπρεπε να ελευθερωθούν από την Αμερικανική κυβέρνηση. Η Διεθνή Αμνηστία επανειλημμένα επέκρινε τι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση αυτών των πέντε φυλακισμένων ε, που ήταν αντίθετο μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα όλοι οι βαθμοί δικαστικοί ολοκλήρωσαν όλε τι δικαστικέ διαδικασίε. Η Κουβανή είναι στη φυλακή 14 χρόνια και εξαρτάται μόνο από τον πρόεδρο Ομπάμα να διορθώσει αυτή την τεράστια αδικία, σοβαρή αδικία. Ζητάμε και από το Ευρωκοινοβούλιο και διακόπτει ο πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε συνάδελφε Βάτιμο. Η συνάδελφο Μιράντα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε η διασφάλιση της βιοπικιλότητα είναι ένας από τους κύριους στόχου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυστυχώ δεν υλοποιούνται πάντα με την αναγκαία αποτελεσματικότητα. Είναι η περίπτωση τη Γαλλικία, όπου έχουμε χιλιάδες εκτάρια που χάθηκαν φέτο, όπου οι πυρκαγιές, οι δασοπυρκαγιές κατέστρεψαν τεράστιες περιοχές ανεκτήμητη βιολογική αξία. Εδώ και ένα μήνα αυτό αυτή είναι μία από τις ε, πτυχές ε, του ε, εθνικού δρυμού που είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης και σήμερα έχει καταστραφεί. Και γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγει πολιτικές πρόληψης των δασοπυρκαγιών. Περιφερειακές πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο να αποφευθεί η εγκατάλειψη της γης από τους γεωργούς και τους καλλιεργητές και θα διασφαλίσει την διασφάλιση, τη διατήρηση αυτών των οικοσυστημάτων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε για το μέλλον μια πράσινη περιοχή στην Ευρώπη εκεί. Θα σε ευχαριστούμε συνάδελφε Μιράντα. Ο συνάδελφος Μάιερ δυστυχώς δεν παρίσταται. Και γι' αυτό θα λάβει τον λόγο τώρα ο συνάδελφος Τσανώνη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. επιστήσω την προσοχή σα σε εκείνο που θα μπορούσε να συμβεί σύντομα σε, μια, σε ένα πιο όμορφα δάση ε, του Κανσίλιου, που είναι μεταξύ Βένετο και Φριούλη τις περιοχές αυτές. Πρόκειται περί περιοχής με πολύ μεγάλη ε, φυσική αξία και ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Αυτό το δάσος ήδη προστατεύεται από την γαλινότατη δημοκρατία της Βενετίας για πρώτη φορά μετά από αγόρευση που χρονολογείται από εκατοντάδες χρόνια θα, ανοίξει, θα επιτραπεί το κυνήγι για χιλιάδες ελάφια από το Μπελούνο, το Τρεβίζο, Βένετο και Φριούλη. Λοιπόν, βαρβάρος θα σκοτωθούν και τα θηλυκά ελάφια, τα έγκυα που είναι έτοιμα να γεννήσουν, Όπω αποφασίστηκε από διάφορα σχέδια φόνου, διότι θεωρείται ότι υπάρχει υπερβολικός Ε, ενώ πολλέ ενώσει το αμφισβητούν. Οι Ιταλικέ αρχέ όμω δίνουν ελεύθερη δίωδο σε, σε αυτούς τους φόνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με μεγαλύτερο, ε, μεγαλύτερη δράση να θέλει να, να εφαρμοστούν οι οδηγίε που στατεύουν την ποικιλότητα και θα πρέπει να εφαρμόσει κυρώσει κυρώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση που παραβαίνει αυτέ τι οδηγίε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Τσανώνη. Η συνάδελφος Τσούμπερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του λαού της Πορτογαλίας επιδεινώνεται σημαντικά. τα επίπεδα διαβίωσης βρίσκονται σε, σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Και αυτό σε σχέση με τη σύμφωνη γνώμη της πορτογαλικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι η πολιτική αυτή ακολουθεί την ορθή κατεύθυνση. Όμως βλέπουμε εδώ την ύφεση, την καταστροφή των θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της καταστροφή θέσεων απασχόλησης πάνω από 200.000 θέσεων. Οι ε, Πορτογάλοι ζουν κάτω από τη φτώχεια. Αυτά όλα τι σημαίνουν, ότι η Πορτογαλία βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση όταν έχουμε την ε, αύξηση, της, ε, της, την μείωση της κατανάλωσης, όταν έχουμε μείωση των εισοδημάτων, όταν έχουμε το πάγωμα των μισθών. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Πορτογαλία βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση και όλα βαίνουν καλώς, όταν έχουμε τις ιδιωτικοποιήσεις, όταν έχουμε την περικοπή κοινωνικών υπηρεσιών και δημόσιων υπηρεσιών και ιδιαίτερα όσον αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση, όλα αυτά τι σημαίνουν, ότι η Πορτογαλία βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε συνάδελφε Σούβερ. Ολοκληρώνονται τώρα οι παρεμβάσεις του ενός λεπτού με την παρέμβαση συναδέλφου Οιουλάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αρχές του Κρεμλίνου προβαίνουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά ε, την απόκτηση 20 εκατομμυρίων αξίας ακινήτων στο Παρίσι για να φτιάξουν μια εκκλησία ε, του, για το Πατριαρχείο, για τον, για τον, Κυριλικό ε, που δεν αρκείται στον ιστορικό καθεδρικό Νεύσκι. οπότε έτσι έχουμε την κατασκευή 200 εκκλησιών σε 10 χρόνια και θέλουν να φτάσουν στα 500, 500 εκκλησίες νομίζω ότι σε κάθε δημοκρατία πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Οπότε είναι καθήκον να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από αυτού του είδους τις θρησκευτικέ δογματικές επιθέσεις του Ορθόδοξου Κρεμλίνου οπότε έτσι θα πρέπει να αποφασίσουμε πρέπει να, ε, να επιτρέψουμε να προβεί σε αυτές τις πράξεις το τόσο αμφίβολο καθεστώ του. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Όγιουλαντ. Η σημερινή μας σε ολοκληρώθηκε εδώ. Η αυριανή θα διεξαχθεί αύριο 18 Απριλίου Τετάρτη από τις 9 ως τις 15.00. Ε, η, η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμη.